Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 9 Uhr. η ώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Έχετε την μέση διάταξη. Το σημείο 1 είναι η έγκριση ημερησία διάταξη. Έχετε προτάσει τροποποίηση ή αντιρρήσει. Εάν όχι, η ημέρησια διάταξη θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Πάμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της 22 Σεπτεμβρίου και 7 η Οκτωβρίου ως ήθιστε εάν μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίασης δεν εγερθεί καμία αντίρρηση τότε θεωρούνται τα πρακτικά ως εγκεκριμένα. Σημείο 3. Ανακοινώσεις. Εξ από σήμερα η συνεδρίασή μας θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο με web streaming και θα βρίσκεται και στα οπτικοακουστικά αρχεία του Κοινοβουλίου. Μόνο από σήμερα. Ε. Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν να έχετε ε, γνώση συγκεκριμένων στοιχείων της αλληλογραφίας μας μπορεί η γραμματεία να σας τα δώσει άλλε, <clears throat> άλλε ανακοινώσεις έχουμε την εμπορική συμφωνία με την Σιγκαπούρη και αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες αλλά αφορά και τις επενδύσεις πλέον συμφωνία αυτή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το σημείο. Κάτι το οποίο μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι ότι η Κομισιόν έχει αποφασίσει να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διακριβώσει πότε μια συμφωνία θεωρείται συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πότε θεωρείται ότι είναι μεικτή μικτού χαρακτήρα συμφωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα κριτήρια τα οποία οδηγούν στον προσδιορισμό μιας συμφωνίας ως μικτής συμφωνίας. Για τον ΠΟΕ έχουμε κάποιες όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικές ειδήσει. 21 Οκτωβρίου Θεωρούσαμε ότι θα υπάρξουν πρόοδοι στη συνεδρία του ΠΟΕ στις 21 Οκτωβρίου, από ό,τι ξέρω όμως δεν υπήρξε απόλυτα, απολύτως καμία πρόοδο σε σχέση με τις λεγόμενες trade facilities, τις διευκολύνσεις εμπορίου, οι οποίες προχωρούν με βήμα σημειωτών, όπως και στο παρελθόν, στον ΠΟΕ. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγματών. Και τον Ιούνιο υπήρξε μια μικρή κίνηση σε ό,τι αφορά το Aid for Trade. Έχουμε τώρα και μια εμπορική διαφωνία, μια διαμάχη με τη Βραζιλία για τη νέα φορολογική δομή του βραζιλιανικού δικαίου που μπορεί να θεωρηθεί ότι ε, πλήττει διακριτικά τις, τα ευρωπαϊκά προϊόντα 18 Νοεμβρίου θα έρθει στην Επιτροπή ε, Διακανονισμού Διαφορών του ΠΟΕ. Στις 9 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Παρόσο με τον πρόεδρο πρόεδρος του Καζακθάνου Αζερμπάιεφ υπέγραψαν μια συμφωνία, μονόγραψαν καλύτερα μια συμφωνία η οποία θα πρέπει και αυτή να μας απασχολήσει και η οποία θα πρέπει να αναλυθεί σε συνδυασμό με την είσοδο του Καζακστάν στον ΠΟΕ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίσης και το θέμα της Δυτικής Αφρικής και της Οικονομικής Ένωσης της ε, Δυτικής Αφρικής. Έχουμε επίσης και με την κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής μια ε, συμφωνία για εταιρική και εμπορική σχέση. Εδώ η Κένια βρίσκεται στο στόχαστρο, η οποία ε, ανήκει στις, ε, στις χώρες οι οποίες ήταν οι λιγότερο ανεπτυγμένες. Τώρα όμως δεν υπάρχει, δεν είναι πια σε αυτή την κατηγορία, επομένως δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια συμφωνία αυτού του είδους και έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα των Φιλιππινών του κατά πόσο μπορούμε να προβούμε σε μια παράταση του καθεστώτος προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων ή όχι. Για μένα δεν είναι το καλύτερο Ε, πρόκειται για το Εκουαδόρ, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος, δεν είναι οι Φιλιππίνες που πρόκειται να παραταθεί η συμφωνία προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων. Έρχομαι στο Κάρι Φόρουμ τώρα, μετά από πέντε χρόνια. Θα πρέπει να επανεξεταστεί η συμφωνία που έχουμε και οι πρώτες συζητήσεις για το θέμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσουν ε, θα γίνουν επί τη βάση μιας μελέτης που θα παρουσιαστεί στις 6 Νοεμβρίου. Κίνα τώρα. Εδώ θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η αντιπαράθεση με την Κίνα σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες έχει εξομαλυνθεί και υπάρχει μια κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας περιλαμβάνει την ε, δήλωση της κινέζικης κυβέρνησης ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει καμία διάκριση στους δημόσιους διαγωνισμούς σε βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επίσης η χρηματοδότηση της ε, έρευνας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θα γίνεται με τρόπο ώστε δεν θα προξενεί στρεβλώσεις. Επομένως έχει ξεπεραστεί αυτή η διαμάχη στην επόμενη συνεδρία μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της παραγωγής κλώστο-εφαντουργικών στο Μπαγκλαντές και τα προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν με την πυρκαγιά και την κατάρρευση ενός κτηρίου που οδήγησε σε πολλούς θανάτους και επομένως θα έχουμε και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σε σχέση με τις εμπορικές προτιμήσεις. Όλα αυτά ήταν οι ανακοινώσεις μου. Πάμε λοιπόν στο σημείο 4 το χρονοδιάγραμμα για τις συνεδριάσεις μας του 2015. Έχετε τις ε, ημερομηνίες οι οποίες προέκυψαν μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τις άλλες επιτροπές για να μπορούμε να καθορίσουμε τις αίθουσε την παρουσία διερμηνέων κτλ. Οι συντονιστές σας έχουν δώσει λοιπόν το σχέδιο αυτό για τις ε, συνεδριάσεις μας του 2015 Παρακαλώ καταγράψτε τα όλα αυτά και να εξασφαλίσετε ότι μπορείτε να είσαστε παρόντες στη συνεδριάση των επιτροπών μας. Σημείο 5 τώρα. Απαλλαγή 2013 σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, η απαλλαγή λοιπόν της Κομισιόν. Και εδώ το ελεκτικό συνέδριο έχει δημοσίευσει μια έκθεση και εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε όπως αποφασίσαμε και βάσει της ε, πάγιας πρακτικής μας αυτός ο οποίος είναι αρμόδιος για το, τα θέματα του προπολογισμού στην Επιτροπή μας είναι αρμόδιος και για το θέμα της ε, απαλλαγής και γι' αυτό δίνω το λόγο με μεγάλη χαρά στο Ράιμερ Μπέγκε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει ήδη αντιμετωπίσει την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την απαλλαγή. Θέλω να εστιάσω μονάχα σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Ελεκτικό Συνέδριο έχει συντάξει μια ειδική έκθεση που αφορά τις προτιμησιακές ε, εμπορικές σχέσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει αποφασίσει να λάβει υπόψη της αυτή την ειδική έκθεση και στη διαδικασία ε, απαλλαγής, οπότε και για μας θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας. Υπάρχουν και μια σειρά από σημεία τα οποία έχει εξετάσει το ελεκτικό συνέδριο, μεταξύ των οποίων το να του ελέγχου των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών των ε, συμφωνιών και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που εφαρμόζονται για το να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στις στους προτιμησιακούς δασμούς ώστε να υπάρξουν προβλήματα, ώστε να μην υπάρξουν συγγνώμη, προβλήματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι η Κομισιόν δεν έχει αναλύσει πλήρως όλες τις οικονομικές συνέπειες των συμφωνιών προτιμησιακής εμπορικής σχέσης. Μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν η έκθεση αντικτύπου και η ποιότητα των αναλύσεων ε, πηγαίνει προς μια πορεία βελτίωσης, αλλά μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Λέει επίσης το ελεγκτικό συνέδριο ότι υπάρχουν ασθενή σημεία στη διαδικασία ελέγχου στα κράτη-μέλη, αλλά επίσης υπάρχουν και σημεία αδυναμίας σε ό,τι αφορά το ρόλο της Κομισιόν και τον έλεγχο τον οποίο πρέπει να εποπτεύει τον έλεγχο των κρατών μερών πρέπει να εποπτεύει η Κομισιόν. Αναφέρεται επίσης ε, ότι στις 3 με 4 ε, Δεκεμβρίου θα υπάρξει συζήτηση με την Κομισιόν ενός ε, σχεδίου χρωμοδότησης. Το ελεγκτικό συνέδριο όπως σας είπα προηγουμένως ζητά μια πιο εντατική αξιολόγηση και ζητά να υπάρξει μια πιο επακριβής ανάλυση του κατά πόσο αυτές οι συμφωνίες προτιμησιακού εμπορικού χαρακτήρα επιτυγχάνουν τον οικονομικό και τον πολιτικό του στόχο και επίσης θέτει το ερώτημα του σε ποιο βαθμό η χρήση αυτών των ε, εμπορικών συμφωνιών μπορεί σε κέριους τομείς να βελτιώσει την ε, οικονομική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποιοι είναι οι πόροι οποίοι προκύπτουν για τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι πρέπει να καταρτήσουμε ένα προφίλ κινδύνου για αυτές τις συμφωνίε, ώστε όλα τα κατημέλη να έχουν μια κοινή βάση για την ανάλυση κινδύνου και για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ζητά από τα κατημέλη να έχουν πιο αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου των κινδύνων και να βελτιώσουν τα συστήματά τους και περιλαμβάνει και ορισμένε προτάσει προ την Κομισιόν, μια σειρά συστάσει προ την Κομισιόν. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, αλλά και εμεί ω Επιτροπή η οποία δίνει γνωμοδότηση θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Στι 3 με 4 Δεκεμβρίου, όπω σα είπα, θα υπάρξει συζήτηση με τα αρμόδια μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Επομένω, μπορούμε να περιμένουμε κάποιε πληροφορίε από τη συνεδρία σε αυτήν. Ένα δεύτερο σημείο, το οποίο είναι επίση σημαντικό και έχει να κάνει με τη διαδικασία του προπολογισμού, το εξή θέμα. Πρόκειται για τα κέντρα επιχειρηματικού χαρακτήρα στην Ινδία, στην Κίνα και στην Ταϊβάν. υπάρχουν τέτοια κέντρα και άλλα κέντρα τα οποία είναι υποσχεδιασμό σε, στις χώρες αυτές και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με την Κομισιόν. Εμείς ζητήσαμε να υπάρξει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του ρόλου αυτών των κέντρων επιχειρηματικού χαρακτήρα και για μας αυτό αποτελεί μια προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την αξιολόγηση προτού υλοποιηθούν αυτά τα κέντρα και θέλουμε να ξέρουμε από την πλευρά της Κομισιόν πότε θα μπορέσει να μας δώσει μια τέτοια έκθεση αξιολόγησης αυτών των επιχειρηματικών κέντρων ώστε να μπορέσουμε ενδεχομένω να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτή τη διαδικασία στη διαδικασία απαλλαγή του 2013. Αυτά είναι τα δύο σημεία στα οποία ήθελα να εστιάσω και είμαι έτοιμο να ακούσω τι προτάσει και τι ε, ιδέε των συναδέλφων. Η αν κατάλαβα καλά, η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να γίνει στις 21-22 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία... Ε, δεν, έχω, δεν έχω γνώση κάποιας ενδεχόμενης ε, διορισμού από τις ομάδες για σκιώδεις συγητές. Γνωρίζει κανείς αν θα, ποιοι θα είναι οι σκιώδεις συγητές. Ρωτάω πρόεδρος στα διάφορα κόμματα, συντηρητική, άλντε, ε, σοσιαλιστές, κανείς δεν ξέρει, Γκούε, ο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Εμείς λοιπόν θα, ε, θα, αναλάβουμε, θα αναλάβω αυτό το θέμα και θα σας παρουσιάσω τις απόψεις μας για τους πράσινους. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα είναι αρμόδιος και η EFTD, η Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία, Εντάξει. Ναι. Αν έχουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, όπως είπε και ο Ράιμερ, θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό, γιατί πράγματι είναι δική μας υπόθεση να αξιολογήσουμε τις εμπορικές συμφωνίες. Μπορώ να δώσω τώρα στην Κομισιόν το λόγο στον κύριο Φανπούκε. Thank you much, uh, Chairman, and thank you uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και κύριε Ισηγητά. Από ό,τι κατάλαβα η συζήτηση της ειδική έκθεσης θα γίνει αρχές Νοεμβρίου, τώρα δηλαδή, και... Όχι, αρχές Δεκεμβρίου, με συγχωρείτε. Και φυσικά θα συμμετάσχουμε και εμείς. Δύο θέματα που έθιξε ο εισηγητής ενδιαφέρουν και εμάς, δηλαδή τα σχόλια του συνεδρίου για τις πιθανές βελτιώσεις. Εμείς συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι πράγματι μπορεί να υπάρξει βελτίωση και έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε βελτιώσεις. Σύμφωνα με τις συστάσεις που αναφέρει ακριβώς η έκθεση του συνεδρίου. Όσο για τα λεγόμενα risk profiles, έχει γίνει νομίζω κάποια αξιολόγηση ήδη που αναλύει τι είδους risk profiles πρέπει να καθοριστούν αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη κανένα. Τώρα για τα επιχειρησιακά κέντρα, business centers, εμείς δεχόμαστε τη συνεργασία που υπάρχει ήδη μεταξύ Κοινοβουλίου και των διαφόρων υπηρεσιών της Κομισιόν και θέλουμε να εξεταστούν από κοινού και σε λεπτομέρεια αυτά τα θέματα. Για τα τρία κέντρα Ταϊλάνδη, Κίνα, Ινδία πρέπει να πούμε ότι έγινε μια μετατόπιση από την εγκαθίδρυση νέων επιχειρησιακών δομών στην στήριξη ευρωπαϊκών δομών. Από ό,τι κατάλαβα όλες οι αξιολογήσεις που έγιναν ε, γνωστοποιήθηκαν και στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και φυσικά τέτοια συνεργασία θα συνεχίσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Μπέγκε, θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Όχι. Ωραία. Το χρονοδιάγραμμα. Θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κύριου Μπέγκε στις 4 Δεκεμβρίου και μετά θα είναι η 11η Δεκεμβρίου η προθεσμία για τις τροπολογίες. 21-22 θα ψηφίσουμε, Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σημείο 6. Η Συμφωνία ε, Προτιμησιακού Εμπορικού Χαρακτήρα με τη Μολδαβία και έχουμε συζητήσει για το θέμα αυτό στα πλαίσια άλλων ήδη ε, θεμάτων. Ο κ. Σόισερ, ο οποίο είναι ο μόνιμο εισηγητή για την Μολδαβία, είναι ο αρμόδιος εισηγητή και του δίνω το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη παρουσίαση των διακευωμένων συζητούμε μια πρόταση της Κομισιόν για να τροποποιήσουμε το καθεστώς των αυτονόμων ε, εμπορικών σχέσεών μας με τη Μολδαβία, που είναι το καθεστώς που ισχύει από το 2005. Πρόκειται για τρία είδη δασμών, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικό χαρακτήρα για την μολδαβική οικονομία, η οποία, όσο γνωρίζετε, είναι κυρίως μια αγροτική οικονομία. Το πλαίσιο όμως είναι ότι το εμπάργκο της Ρωσίας για τα αγροτικά προϊόντα της Μολδαβίας που εισήχθη ετέθησε ισχύ στις 21 ε, Σεπτεμβρίου και εμείς πληττόμεθα από αυτό το σύστημα. Πρόκειται εδώ για τα, την εισαγωγή μήλων, 40.000 τόνοι, επιτραπέζια σταφύλια 10.000 τόνοι και επίσης ε, δαμάσκηνα 10.000 τόνοι. Είναι φυσικά ίσονες ποσότητες σε σχέση με, τις, ε, με την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 0,4% της ευρωπαϊκής παραγωγής είναι τα μήλα, 0,6% τα σταφύλια και 0,7% τα δαμάσκηνα. Επομένω είναι συμβολικές ποσότητες για μας, για την μολδαβική οικονομία όμως και την παραγωγή φρούτων και λαχανικών όπου απασχολούνται 250.000 άτομα που εργάζονται κυρίως σε πολύ μικρά αγροτεμάχια. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο υποστήριξης της οικονομίας τους και τους δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσουν σε οικονομικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που ελοχεύουν για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτα αμεληταίοι για πολλούς λόγους για λόγους γειτονία και για λόγους πολιτιστικούς όλα αυτά τα προϊόντα θα πάνε μονάχα στην αγορά της Ρουμανίας. Μόνο για τα μήλα υπάρχει κάποια ευαισθησία, γιατί φέτος είναι ένα ευαίσθητο προϊόν. Σε ό,τι αφορά όμως την ποιότητα και την... το επίπεδο εξέλιξης των μεθόδων συσκευασίας και εμπορίας, είναι απίθανο ότι τα μήλα αυτά της Μολδαβίας τα οποία θα θεωρηθούν στη Γαλλία και την Ιταλία κατά πάσα πιθανότητα ως βιομηχανικά μήλα και θα συναγορίζονται τα εγχώρια εκεί μήλα. Τα περισσότερα από αυτά θα βγουν στην αγορά της Ρουμανίας η οποία εφέτος θα μπορέσει να απορροφήσει όλα αυτά τα προϊόντα λόγω των ευνοϊκών συνθήκων η ρουμανική παραγωγή θα είναι 22% υποδέστερη από την περσινή και η ποσότητα αυτή που αναφέρουμε είναι το 8% της παραγωγής της Ρουμανίας η οποία μπορεί να απορροφήσει όλη τη μολδαβική παραγωγή και να έχει ακόμα περιθώριο 14% για να εισαγάγει μήλα από αλλού. Δεν υπάρχει απώλεια εισοδήματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί <clears throat> δεν υπάρχουν ε, μήλα ή άλλα ε, φρούτα και λαχανικά που να μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά με χαμηλότερη τιμή από την τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα υπάρξει λοιπόν απώλεια εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι υπάρχουν πιο πολλά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αν θέλουν οι συνάδελφοι λεπτομέρειες, αλλά γενικά μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος μπορεί να γίνει εύκολα <clears throat> αποδεκτός από εμά και συγχρόνως θα βοηθήσει ιδιαίτερα τη μολδαβική οικονομία όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εργάζονται στον τομέα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω σε όλου όλους τους συναδέλφους <clears throat> να αποδεχτούν την πρόταση της Κομισιόν χωρίς καμία τροποποίηση. Και η πρόταση επίσης δημιουργεί για ορισμένου ανησυχίες επειδή υπάρχουν κάποιες ε, τροποποίησεις των εμπορικών κωδίκων σε αυτή την ε, πρόταση, οι οποίοι έλκονται από τη μεταρρύθμιση του τελωνιακού κώδικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρσι, αλλά εγώ έχω ελέξει και πραγματικά δεν υπάρχει καμία απολύτως εμπίπτωση. είναι μια μικρή τεχνική προσαρμογή και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ κύριο Σβίνκλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ ε, πολύ για την παρουσίαση. Ε, πολύ εμπεριστατωμένη. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε πολλά πράγματα. Ε, ως εκπρόσωπος τώρα του ΕΛΚ ε, εμείς συμφωνούμε να δοθούν εμπορικές προτιμήσεις στη Μολδόβα έχουμε συχνές επαφές ε, προγραμματισμένες μέσω της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για τη, με τη Μολδόβα αλλά στην ουσία μιλάμε για τη Ρωσία αν δει κανείς πίσω από τα από τη βασική σελίδα η Γροσία είναι το πρόβλημα και το εμπάργο που επέβαλε στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Είμαι πολύ περήφανος που η ΙΝΤΑ, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, είναι, έχει δραστηριοποιηθεί πολύ για αυτό το θέμα και που γιατί το εμπόριο είναι πραγματικά αποτελεί πραγματικά μια πρακτική βοήθεια για τους εταίρους μας της ε, ε πολιτικής γειτονίας και η προτιμησιακή αυτή κατάσταση ε, ισχύει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου του τρέχοντος έτους και βεβαίως θα εκπνεύσει στη 2015 όταν θα εκπνεύσει και το καθεστώς ε, που έχουμε ε, με την Μολδόβα. Είναι επίγουσα η κατάσταση, δείχνουμε πολιτική εδώ ηγετική στάση και Εάν γίνει δεκτός αυτός ο φάκελος θα είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ προτείνω να εγκρίνουμε την πρόταση της Κομισιόν χωρίς τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσάντελ δεν είναι εδώ, ο κύριος Ρεν είναι εδώ. Ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, κύριο Σόλτς. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση της έκθεσης και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει χωρίς καμία τροποποίηση να εγκρίνουμε την ε, πρόταση αυτή. Μία μικρή παρατήρηση μονάχα. Είπε ήδη ο κύριος Βίνκλερ ότι φυσικά υπάρχει το θέμα των σχέσεων με την Ρωσική Ομοσπονδία και υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Μολδαβίας και εδώ θα πρέπει να δούμε το συνολικό πλέγμα των εμπορικών σχέσεων και η δική μου <clears throat> επιθυμία θα ήταν όταν συζητήσουμε για την πραγματική εφαρμογή αυτής της εμπορικής συμφωνίας να μην ε, έχουμε την ε, να μην θέσουμε εμπόρια και για μεταποιημένα προϊόντα γιατί τα επιτραπέζια σταφύλια της, της Μολδαβίας μπορεί να είναι βασική πρώτη ύλη και για την παραγωγή ίνου σε άλλες χώρες. Να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτά τα προϊόντα μπορούν να έχουν χρήση μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά για στόχο της μεταποίησης. Λοιπόν, πρέπει να τα ελέγξουμε όλα αυτά, λέει ο πρόεδρος. Ο Ζαντό δεν είναι εδώ παρόν και έχει το λόγο τώρα η κυρία Λεπέν. Η Συμφωνία Σύνδεσης Ένωσης Μολδαβίας εξαιρεί τα αγροτικά προϊόντα, λέει το κείμενο. Η Μολδαβία ενέκρινε ένα φιλόδοξο πολιτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και πλησιάσματος οικονομικού με την Ένωση. Σε μερικά χρόνια λοιπόν μπορεί να γίνει μέλος της Ένωσης, αυτό ελπίζεται τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος, στο μακρύ κατάλογο που δείχνει την ε, κατάσχετη όρεξή σας. Παρ' όλα αυτά εφευλήθηκε εμπάργκο στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Μολδαβία και παράλληλα ζητάτε από τους κοινοβουλευτικούς να αυξηθεί την ποσόστοση εισαγωγών μήλων από τη Μολδαβία. Επομένως όλοι οι γεωργοί της Ένωσης πρέπει να αφήσουν χώρο για τα προϊόντα της Μολδαβίας στις αγορές τους, ενώ η αγορά των οποροκυπευτικών έχει σχεδόν καταστραφεί μετά από το ρωσικό εμπάρκο και μετά από τη σύναψη και άλλων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με σκοπό την αύξηση του αθέμητου ανταγωνισμού. Έτσι, δεν μας λέτε ούτε μια λέξη για τις δυσκολίες των Γεωργών, ούτε μια λέξη κάθε δύο μέρες περίπου ένας γεωργός αυτοκτονεί στη Γαλλία. Κάθε δύο μέρες αυτοκτονεί ένας γεωργός στη Γαλλία γιατί δεν καταφέρνει πια να ζήσει από τη δουλειά του. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, με με τη Μολδαβία, τίνεται μερικά ψίχουλα και τίποτα δεν βελτιώνεται. Σήμερα γίνεται μια σημαντική απεργία γεωργών σε όλη τη Γαλλία που καταδικάζει την πτώση των ε, τιμών των αγροτικών προϊόντων μετά από το ρωσικό εμπάργκο. Κύριοι Ευρωπαϊστέ, θα θέλατε όλοι οι πολίτες του κόσμου όπως λέτε ή οι κοσμοπολίτες ε, να αγαπάτε όλους τους πολίτες του κόσμου αλλά δεν αγαπάτε τους πολίτες τους δικούς σας. Δεν σας αφορά η καταστροφή αυτή της αγοράς των αγροτικών προϊόντων μετά από το ρωσικό εμπάρκο. Θέλετε συνεχώς μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών. Ενώ δεν είναι προς το συμφέρον ούτε ημών ούτε των Μολδαβών. Η ιδεολογία σας σας το επιβάλλει αυτό και εγώ είμαι κατά τα Εντάξει, θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Ντλουκ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Δύο πράγματα. Νομίζω πως ο εισηγητής έχει πει τα βασικά και έπειτα να μιλήσω για το πλαίσιο και μετά για το περιεχόμενο της πρότασης. Ε, όσον αφορά το πλαίσιο έχουμε όντως δει όπως η Ρωσία επιβάλλει διάφορα εμπάργκο στην ε, Μολδαβία και αντίθετα με τα όσα είπε η κυρία Λεπέν αυτό δεν ε, είναι συνέπεια του ευρωπαϊκού εμπάργου αλλά είχαν επιβληθεί αυτά προηγούμενα. Μάλιστα ξεκίνησαν ε, λίγο μετά την ονειροστικοποίηση της συμφωνίας ε, με τη Μολδαβία. Ε, ε υπήρξε εμπάργο τον Ιούλιο για το κατεργασμένο κρέας, έπειτα για τα, ε, τις κονσέρβες φρούτων και τα λαχανικά και έπειτα η Ρωσία αφαίρεσε την ε, τις προτιμησιακές, τα προτιμησιακά τέλη για τις εισαγωγές από τη Μολδαβία που κάλυπταν 16% των εξαγωγών της Μολδόβας από, προς τη Ρωσία. Ε, οι απώλειες είναι 130 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ε, λόγω του εμπάργου. Η Ρώσα στόχευσε πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα τα οποία μαζικά εξάγονταν προς ε, την ίδια και ε, Φυσικά δεν χρειάζεται να τονίσουμε τις πολιτικές συνέπειες όλων αυτών για τις επερχόμενες εκλογές στην Μολδόβα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργό Ιάνκα ζήτησε από τον Πρόεδρο Μπαρόζο τον Ιούλιο του 2014 να ε, υπάρξει αυτή η συμφωνία. Για τα τρία αυτά προϊόντα τώρα, μήλα, στα σταφύλι και δαμάσκηνα και για τα ανευτελών προϊόντα, τα duty προϊόντα, τα οποία μπορούν να μπαίνουν στην Ένωση. Έχουμε και ένα ακόμα στοιχείο σημαντικό που είναι βέβαια προσωρινό μέτρο θα εκπνεύσει με την εκπνοή της ε, ισχύουσα αυτόνομης ε, μπορική προτίμησης, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2015. Όσον αφορά τα προϊόντα και τις ποσότητες για τις οποίες ε, προτείνεται το μέτρο, ε, πρόκειται για εξαιρετικά μικρές ποσότητες σε σχέση με την ευρωπαϊκή παραγωγή, γιατί μιλάμε για 0,8% της μολδαβικής παραγωγής σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή παραγωγή, 1,4% για τα δαμάσκηνα και ένα και ένα αντίστοιχο ποσοστό για τα επιτραπέζια στα φύλλα. Ε, όμως θα έχει μεγάλο ωφέλη για τους Μολδαβούς παραγωγούς. Ευχαριστώ. Μπορώ να ξαναδώσω στον εισηγητή πάλι το λόγο στον κύριο Ναι. Να σας ξανααναφέρω κάποια επιχειρήματα στα γαλλικά. Για να διευκρινίσω με μεγαλύτερη σαφήνεια τα όσα είπα και προσχάριν της κυρίας Λεπέν. Αν κάποιος εκμεταλλεύεται τον πόνο των Γάλλων γεωργών, Σίγουρα δεν είναι οι κατακαημένοι Μολδαβοί που θα ε, κερδίσουν λίγο από τα μέτρα που προτείνουμε και ελπίζουμε θα εγκριθούν σε λίγες εβδομάδες. Ήδη εξήγησα ότι η ρουμανική παραγωγή φέτος έπεσε κατά 22%. Το κομμάτι το οποίο προτείνουμε εδώ είναι 8% της ρουμάνικης παραγωγής. Ε, υπάρχει μια μικρή διαφορά στις στατιστικές που έχω εγώ με τα, σε σχέση με το όσο μας είπε η Κομισιόν. Το όσο, αυτά που προτείνουμε εμείς, 40.000 τόνοι, είναι 0,4% της ευρωπαϊκής παραγωγής, ενώ το σημερινό αυτό τμήμα η ποσόστοση και της ε, συμφωνίας ε, της ελεύθερων συναλλαγών που είναι παρόμοιο αξίζει 0,8% είναι αλήθεια. Αλλά σήμερα μιλάμε τις 40.000 τόνους των αυτόνομων μέτρων. Τώρα, από την άποψη της ποιότητας είναι προφανές πως αυτά τα προϊόντα που θεωρούνται βιομηχανικά στην ουσία βιομηχανικά στη Γαλλία και στην Ιταλία ποτέ δεν θα έρθουν σε ε, ανταγωνισμό με τα Ιταλικά και Γαλλικά προϊόντα. Τώρα, αν θέλουμε να συγκρίνουμε αυτήν την, το δράμα που ζει ο γεωργικός τομέας της Γαλλίας με το μικρό αυτό πως όγκο φρούτων που θα καταναλώσει η ρουμανική αγορά φέτος πραγματικά είναι κάτι πολύ φτηνό και άτιμο. Δεν υπάρχει λόγος να παίζουμε έτσι με τον πόνο των λαών. Ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 11η Νοεμβρίου στις 6 η ώρα το απόγευμα. Στις 3 Δεκεμβρίου θα συζητήσουμε και πάλι για τις τροπολογίες και στις 4 Δεκεμβρίου μετά θα γίνει η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται να γίνει ίσως το Δεκέμβριο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουάριο 2015. Σας ευχαριστώ πολύ και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 7. Πρόκειται για τα μέτρα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα σταθεροποίησης της διαδικασίας ε, προσχώρησης και εδώ αφορά την Βοσνία Ζεγοβίνη το σύνολο αυτών των μέτρων. Έχουμε εδώ ορισμένε ε, δυσκολίες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να εξετάσουμε γενικά τη συνολική διαδικασία έναντι των Δυτικών Βαλκανίων. σε ό,τι αφορά τα εμπορικά θέματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και δίνω λοιπόν ευχαριστώ στο λόγο στον εισηγητή, του κύριο Μπετίνη. cari colleghi, rappresentanti della Commissione. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι της ε, Κομισιόν, πρέσβης της Δημοκρατίας της Βοσνίας, ε, σήμερα ε, ξεκινά η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας για την οποία είμαι εισηγητής που προέβλεπε ένα ειδικό προτιμησιακό καθεστώς για τη Βοσνία όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές. Στόχος μου είναι να ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή την γνώμη όλων των βουλευτών της Επιτροπής ΙΝΤΑ, καθώς και να, να εμβαθύνουμε σε κάθε συγκεκριμένη πτυχή της απόφασης και την αιτιολόγηση αυτής, όπως την υποβάλλει η Κομισιόν στην, στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις ικανότητες ε, καθώς και τα επιχειρήματα των διαφόρων ε, βοσνίων εκπροσώπων ε, ξεκινώντας από τον πρέσβη στις Βρυξέλλες. Προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη των εργασιών μας και το υποβάλλω σε συζήτηση. Σήμερα υπάρχει μια, γίνεται η πρώτη πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Στις 20-21 Ιανουαρίου θα μπορούσαμε να, ε, να συζητήσουμε στην Επιτροπή Ίντα για το σχέδιο κανονισμού. Στις 28 Ιανουαρίου προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Τον Ιανουάριο θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε ε, μάλλον να κάνουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες που θα έχουν υποβληθεί και τον ίδιο πάλι το Φεβρουάριο να γίνει και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ίντα για τον οριστικό προπολογισμό και τέλος ολομέλεια του Στρασβούργου για έγκρισή του. Τώρα θα ήθελα μόνο να σας αναφέρω κάποιες αρχικές μου σκέψεις ε, που στην ουσία είναι ανοιχτά ερωτήματα. Η απόφαση που πρέπει να λάβουμε είναι πολύ πολύ λεπτή, γιατί πρόκειται για μια χώρα σε στρατηγική περιοχή που μετά από ένα σωρό τραγωδίες αναζητεί το μέλλον της σε μια σχέση όλα ένα και πιο ολοκληρωμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής, η Βοσνία δυστυχώς έχει μείνει πίσω. Ε, με δυσκολία γίνονται μεταρρυθμίσεις οικονομικές, ε, διοικητικές, οικονομικές, δημοκρατικές που είναι απαραίτητες για να μπορέσει να μπει η χώρα στην Ένωση. Υπάρχει και μια σύγχυση όσον αφορά την, την ηγεσία της χώρας που καθορίζει και την αβεβαιότητα της ε, ε, συζήτησης ε, με τους διεθνούς, διεθνείς θεσμούς. Ωστόσο, όπως είπε πρώτα ο Φίλε και μετά ο Χάν, ε, επίτροποι για τη διεύρυνση, θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με στένος το πορεία της Βοσνίας προς την Ευρώπη. Τόσο μάλιστα που στηρίξαμε τη χώρα με άμεσες ενισχύσεις, ιδιαίτερα για να μπορέσει να βγει από την τραγωδία των πλημμυρών που τη χτύπησε τα τελευταία χρόνια. Με αυτόνομη και μονομερή απόφαση εφαρμόσαμε ένα συμμετρικό και προτιμησιακό καθεστώς ε, για τις εμπορικές μας σχέσεις με την ελόγω χώρα. Εξάλλου το 85% του βοσνιακού πληθυσμού δηλώνει ότι θέλει θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Δεν είχαμε το χρόνο να... Ε, ε, μάλλον θα πρέπει να έχουμε το χρόνο να εξετάσουμε ε, το γεγονός ότι η Βοσνία με την είσοδο της Κροατίας στην Ένωση που οφείλεται στην πολύ σοβαρή δουλειά από πλευρά της χώρας αυτής θα πρέπει να δούμε ωστόσο ταυτόχρονα τις ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών με βάση την πρόταση της Κομισιόν και ε, το, τα όσα έχουν συμφωνήσει οι χώρες των Δυτικών Βαλγανίων μαζί της όσον αφορά το εμπόριο. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το αν θα λήξει το προτιμησιακό καθεστώς για την 1η Ιανουαρίου και για όλες τις χώρες όμως των Βαλκανίων προβλέπεται να παραταθεί μέχρι το 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, αν ανασταλούν αυτά τα αυτόνομα μέτρα, η Βοσνία θα υποστεί μια ζημιά 2.400.000 ευρώ ετησίως. Προφανώς ένα τέτοιο με τον μονομερές μέτρο προ ε, μια χώρα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στηρίξει και να παροτρύνει στις ε, προσπάθειες προσαρμογής στις παραμέτρους ε, της προσχώρησης στην Ένωση θα ήταν παράξενο. Θα πρέπει λοιπόν η Ένωση να προβεί σε όλη την εξέταση του θέματος. Ας πούμε, ε, ένα ρεαλιστικό, μια ρεαλιστική ε, μελέτη για τις ζημιές που θα μπορούσε να υποστεί η Βοσνία εάν δεχτεί την προσαρμογή. Ε, ξέρουμε ότι από αυτού οι εκπρόσωποι της χώρας μιλούν για 33.000 κόσμο που θα χάνε τη δουλειά του. Σας καλώ λοιπόν όλους να εργαστούμε με νυφαλιότητα επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν και γνωρίζοντας ότι φέρουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στην Κομισιόν όχι στον κύριο Λουκρίνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομος γιατί ο εισηγητής τα είπε όλα. Πράγματι εδώ πρόκειται για την πρόταση αν δεν απατώμε, που παρατείνει τις προτιμήσεις από το 11-15 μέχρι το 20. Επίσης είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αντίθετα από τον κανονισμό για τις προτιμήσεις με την Ουκρανία που τις έχετε συζητήσει δεόντως Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για δυνατότητα παγώματος της ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Υπάρχει λοιπόν η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κανονισμό 12-15 και με αυτήν τη ρήτρα μπορούν να ληφθούν μέτρα εφόσον διαπιστωθεί βασική ουσιαστική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν έχει δεχτεί την προσαρμογή της υπάρχουσας συμφωνίας ώστε να ληφθεί υπόψη το προτιμησιακό εμπόριο μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας καθώς και τις συμφωνίες ΕΖΕΣ για την Κεντρική Ευρώπη που ίσχυαν μέχρι την ένταξη της Κροατίας το 2013. Μόνο λοιπόν αν η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεχτεί την προσαρμογή αυτή, μόνο τότε θα μπορέσουν οι προτιμήσεις για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να αρθούν το 16. Μόλις υπογραφεί τέτοια συμφωνία θα έρθουν. Θα επανέλθουμε μάλλον. Αυτό το θεωρούμε ως κίνητρο για το σεβασμό βασικών αρχών της Ένωσης, δηλαδή ότι οι προτιμήσεις που χορηγούμε μόνο μερός αυτόνομα σε τρίτες χώρες δεν, τους επιτρέπουν, δεν τις επιτρέπουν να επιλέξουν με ποιες χώρες μέλη θέλουν να εφαρμόσουν τις προτιμησιακές αυτές εμπορικές σχέσεις. Ελπίζουμε λοιπόν η Βοσνία Ρεσεγοβίνη να επανέλθει σε επικοδομητικές συνεννοήσεις με την Κομισιόν για την προσαρμογή αυτής της ε, συνθήκης και τότε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μήπως μπορείτε να πείτε κύριε κάτι Ντεβίνιε για την κατάσταση εν γέννη πώς είναι η κατάσταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών της, ε, των Δυτικών Βαλκανίων σε σχέση με τα εμπορικά θέματα. you talking about, uh, Αναφέρεστε σε αριθμητικά στοιχεία ή σε προτιμήσεις. Το γενικό πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων με τα Δυτικά Βαλκάνια, τα πράγματα πηγαίνουν καλά ή όχι. Έχετε μιλήσει για την Βοσνία Ζεγοβίνη αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Um, Έχουμε πράγματι κάποιες σχέσεις με ορισμένες από τις χώρες της περιοχής. Βέβαια, δεν είναι τέτοιου είδους ώστε, ώστε θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία τροποποίηση των εμπορικών μας προτιμήσεων. Αλλά βέβαια είναι σχετικά ίσον το εμπόριο με τις χώρες αυτές από την έποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως 1%, 2% του εξωτερικού μας εμπορίου εν συνόλο. Δεν έχω να πω λοιπόν πολλά σε αυτό το επίπεδο, αλλά ε, αν θέλετε να έχετε μια συζήτηση <clears throat> χωριστά για κάθε χώρα της περιοχής, μπορούμε να έρθουμε <clears throat> με συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τα προβλήματα, αλλά δεν έχουμε γενικά προβλήματα με αυτές τις χώρες. Ε, εντάξει, μπορείτε να προετοιμαστείτε ίσως καλύτερα για την επόμενη συνάντησή μας ε, στις 21-22 Ιανουαρίου, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια σφαιρικότερη εικόνα για τις εμπορικέ μας σχέσεις με τις άλλες χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Έρχομαι στους σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Στίαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. και εγώ θα ακολουθήσω την γραμμή που αναφέρατε εσείς κύριε Πρόεδρε, να έχουμε πρώτα μια γενικότερη εικόνα και μετά να εστιάσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι σωστά είπε η Κομισιόν ότι το σημείο εκκίνησης για αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να είναι η ιδέα ότι αυτός ο κανονισμός είναι μια επέκταση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή θα πρέπει να είναι η οδηγός φιλοσοφία της πρότασης ότι θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση των ε, εμπορικών προτιμήσεων και να δώσουμε με τον τρόπο αυτό στις χώρες αυτές τις δυνατότητες να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά με την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένε χώρες οι οποίες εμπίπτουν σε προγράμματα σταθεροποίησης και εταιρική σχέσης θα πρέπει να τροποποιήσουν τις συμφωνίες που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουν υπόψη την νέα αυτή κατάσταση. Είναι πάντα μια δύσκολη απόφαση. Υπάρχει πάντα ο πειρασμός ε, του να είναι κανείς επιλεκτικός, όπως είπε και η Κομισιόν. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και στο παρελθόν. Είδαμε τι έγινε με τους προηγούμενους γύρους ε, διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία, παραδείγματο χάρη, είχε τον πειρασμό στο παρελθόν να διαλέξει μεταξύ Σλοβα... Σλοβα... Σλοβενία και Ουγγαρία κτλ. Αλλά από τότε που η Σλοβενία και η Ουγγαρία έγιναν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα η Κροατία είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια επιλεκτική αντιμετώπιση. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Σερβία η οποία έχει και αυτή κάποια προβλήματα, συμφώνησε και όλες οι άλλες χώρες της περιοχής. Η μόνη χώρα η οποία παραμένει είναι η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη και γι' αυτό συζητούμε. Για αυτήν. Αυτό είναι λοιπόν το γενικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται όλα αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε κάποια ενθάρρυνση στις διαπραγματεύσεις αυτές. Μας δίνει με αυτόν τον τρόπο ένα χρόνο καιρό γιατί <clears throat> ξέρετε ότι τον Οκτώβριο θα λάβουν χώρα εκλογέ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα δώσει λοιπόν αυτό το μέτρο χρόνο στις νέες αρχές εκεί να ξεκινήσουν από την αρχή της ε, διαπραγματεύσεως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να λάβουν υπόψη <clears throat> το γεγονός ότι η Κροατία έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να προσαρμόσουν την αντίστοιχη συμφωνία. <clears throat> Μια τελική παρατήρηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει, όχι βέβαια με την ψήφο του σε ένα κανονισμό, αλλά με ένα ψήφισμα για την πρόοδο της Βοσνίας Αζεγοβίνης στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χάρη στην, ε, σε μια τροπολογία του Τονίνο Πίτσουλα από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, τη θέση του, επομένως, ο κανονισμό αυτός ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη θέση που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> στις αρχές του 2014 στο ψήφισμά του για την ε, κατάσταση προόδου της Βοσνίας στον δρόμο για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μέτρα και φυσικά υποστηρίζω το να υπάρξει μια συζήτηση σε μεγαλύτερο βάθος και μια ανταλλαγή απόψεων όπως έχει προταθεί από τον αρμόδιο εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Οι συντηρητικοί δεν έχουν κάποιον εισηγητή. Η Μαρίκη εφόσον λείπει όλοι, Ρεν. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμβάλει στη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν. Πρέπει οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν και πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για τις διαπραγματεύσεις, αλλά μας ενδιαφέρει επίσης η Βοσνία Ζεγοβίνη να κατανοήσει ότι πρέπει να γίνουν τεχνικές προσαρμογές στις ε, συμφωνίες αυτού του είδους και η Βοσνία δεν μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή τη διαδικασία και άλλες χώρες έχουν ε, αναγκαστεί να προσαρμοστούν με αυτή την τεχνική διαδικασία. Χρειάζεται να συνεχίσει ο διάλογο για να προχωρήσουμε και ο διάλογο δεν είναι μονάχα για τα εμπορικά θέματα. Υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν σε σχέση με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπου πρέπει η Βοσνία Ζεγοβίνη να επιτύχει πρόοδο για να μπορέσει να προσαρμοστεί στη, στα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώ λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πρέπει να είναι σαφέ σε όλου ότι έχει επιβάλει η Βοσνία δασμούσε προϊόντα από την Κροατία. Αυτό όμως δεν συνάδει με το πνεύμα του ελεύθερου εμπορίου σε διμερές επίπεδο και δημιουργεί προβλήματα για τη δημιουργία μια περιοχή ελευθέρου εμπορίου όπω επιθυμούμε και επίση σημαίνει ότι οι καταναλωτέ στη Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει να πληρώσουν υψηλότερε τιμέ για προϊόντα τα οποία εισάγονται από την Κροατία. Για του λόγου αυτού, εγώ υποστηρίζω τη θέση αυτών οι οποίοι έχουν εκφράσει την ε, ελπίδα ότι μπορεί να εξευρεθεί μια λύση το ταχύτερο δυνατό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επίσης χαιρετίζω την ε, συμπερίληψη ρητρών και προνοιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συμφωνία αυτή. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν αντιμετωπίζουμε αυτέ τι προκλήσει και τα τεχνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φέρουν όλε τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η οπτική γωνία δεν πρέπει να απολεστεί από τα όματά μα. Πρέπει όλε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων να συνεργάζονται προ την κατεύθυνση ενό κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος και όχι να παραμείνουν στο παρελθόν τους, το οποίο είναι γεμάτο με τραύματα βέβαια, αλλά θα τις κρατήσουμε μονομένες. Και πρέπει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε μια δυνατότητα στις χώρες αυτές να έχουν μια προοπτική και γι' αυτό ελπίζω ότι η κυβέρνηση της Βοσνίας Ζεχοβίνης θα λάβει υπόψη τις ε, συστάσεις μας και θα τηρήσει τα συμπεφωνημένα. <clears throat> Ευχαριστώ, λέω Από την ΚΟΓΟΕ δεν υπάρχει κάποιος εισηγητής. Έρχομαι στους πράσινους τώρα. Ευχαριστώ κύριε. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση του. Εκτός από αυτά που ήδη υπόθηκαν, υποστηρίζουμε την άποψή σας ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα σφαιρικά και να λάβουμε υπόψη μας τη γενικότερη εικόνα της κατάστασης στα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως ξέρετε, ένα από τα κύρια προγράμματα, ένα από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής μας είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών και κοινωνικών. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω την ανάγκη να γίνεται σεβαστή, να περιλαμβάνεται η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε φορά, αλλά να λάβουμε και την πραγματικότητα υπόψη μας στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου δεν υπάρχει παράδοση σεβασμού της ένομης τάξεως και διάφορα άλλα τέτοια προβλήματα ανάλογα και αφού τονίσουμε λοιπόν τη στήριξή μας για τη ρήτρα αυτή θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή υπάρχει καμία ανησυχία για αυτό το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει καμία περίπτωση γνωστή έχει καμιά πληροφόρηση να μας κάνει από αυτού. Ευχαριστώ τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων θα ήθελα να ζητήσω μάλλον από τις πολιτικές ομάδες όταν παίρνουν το λόγο σκιώδεις όταν υπάρχουν σκιώδεις εισηγητές να μας το λένε για να μπορούμε να τους δίνουμε το λόγο εξ ονόματος της ομάδας των για τους πράσινους τώρα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε εγώ θα είμαι πολύ σύντομος τα βασικά αναφέρθηκαν εμείς συμφωνούμε με όσα ακούστηκαν και ευχαριστούμε θερμά τον εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ. Η ομάδα FDD, Ελευθερία Δημοκρατία, δεν έχουν σκιώδη εισηγητή, άρα δεν υπάρχει κανείς άλλος που να λάβει το λόγο. Μεταξύ μας βρίσκεται και ο πρέσβης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ο κύριος Ίγκορ Νταβίντοβιτς. Νομίζω ότι άκουσε και αυτός τις προτάσεις. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση. Δυστυχώς μάλλον είχε προσκληθεί ο πρέσβης αλλά δεν προσήλθε αυτό. Άρα δεν θα, λάβει κανείς το λόγο εξ ονόματος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να έρθει ο Πεζοχτής σήμερα, αλλά ίσως στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε για το θέμα αυτό να γίνει αυτό δυνατό. Έχει αναφέρει ο εισηγητής τις χρονικές στιγμές. 20 και 21 Ιανουαρίου θα γίνει συζήτηση και μετά μέχρι τις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει να κατατεθούν οι τροπολογίες και τον Φεβρουάριο του 2015, εάν θέλει ο Θεός, θα ψηφίσουμε ή ίσως και το Μάτιο Κύριε Μπετίνη, θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο? Όχι. Νομίζω πως ε, σαφώς εκφράστηκαν οι πολιτικές θέσεις των ομάδων. Φυσικά, ωστόσο, δεν θα ε, πρέπει αυτό να εμποδίσει την εμβάθυνση σε μια ανοιχτή συζήτηση στη διάρκεια των εργασιών μας, ενώ ε, κάποιοι άλλοι υπογράμμισαν και του ευχαριστώ υπογράμμισαν την συμφωνία τους με την θέση της σύντομης με αυτής έκθεσης. Τώρα, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι το μόνο ερώτημα που μου ετέθη, θα ήθελα να πω το εξή. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν στοιχεία για να πούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση, επικρατεί μια κατάσταση υποτίμησης ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, γενικευμένη. Το θέμα το οποίο όμως είναι πολύ λεπτό γιατί αναφέρεται συγκεκριμένα στην αδυναμία ε, ορισμένων, μάλλον ενός από τους υποψηφίους για την Προεδρία του Σέντιτ Φίντσι να μπορέσει να θέσει την υποψηφιότητά του καν για λόγους ενός συνταγματικού άρθρου της Βοσνίας που, που επιτρέπει στις τρεις εθνότητες που συναποτελούν τους πολίτες της Βοσνίας να συμμετέχουν. Φυσικά αυτό είναι δικαίωμα γι' αυτόν, είναι πολύ σημαντικό δικαίωμα που σε μια δημοκρατία πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως. Ε, όσον αφορά λοιπόν το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω πως για τη Βοσνία κυρίως αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα που αφορά και το ίδιο το Σύνταγμα της Βοσνίας και όχι μια γενικευμένη κατάσταση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν πρόκειται δηλαδή για ζημιά ή πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ για τις παρατήρησεις σας. <clears throat> Μας παρουσιάσατε το χρονοδιάγραμμα. Απλώς παρακαλώ την Κομισιόν στην επόμενη συζήτηση να μπορεί να μας παρουσιάσει εν τα εμπορικά θέματα με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και επίσης επαναλαμβάνεται η πρόσκληση στον πρεσβευτή της Βοσνίας Εζεγοβίνης γιατί εμείς θέλουμε και επιζητούμε το διάλογο. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν το σημείο 7 και να περάσουμε στο σημείο 8. Πρόκειται για ένα προσφυλές θέμα για μας, τον έλεγχο ε, εξαγωγών προϊόντων διτής χρήσης και στην τελευταία θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε μια μεταρρύθμιση των κανόνων για τα προϊόντα διτής χρήσης και αυτό έφερε σημαντικά αποτελέσματα γιατί επιφέραμε όχι μονάχα τεχνικές προσαρμογές της νομοθεσίας αλλά θέσαμε και πολιτικές ε, αρχές σε ό,τι αφορά την έκταση του ελέγχου για τα αγαθά αυτά και μετά την Αραβική Άνοιξη είναι σαφές πια ότι προϊόντα διτής χρήσης από την Ευρώπη έχουν χρησιμοποιηθεί για κατασταλτικούς λόγους στις χώρες αυτές. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε ένα καθεστώς εξαγωγών για τέτοια προϊόντα, <clears throat> ώστε η αδειοδότηση των προϊόντων αυτών δεν θα πρέπει να αφορά την δυνατότητα χρήσης του σε άλλες χώρες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο νομικό πλαίσιο και η Κομισιόν μας έχει υποσχεθεί να κάνει μια τέτοια πρόταση. Μέχρι στιγμής δεν έχει όμως διατυπώσει μια τέτοια πρόταση και γι' αυτό οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ζητήσει να υπάρξει ένα ψήφισμα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν για να μας υποβάλει αυτές τις νέες προτάσεις. Και ιδίως εν ώψη της ε, αύξησης της χρήσης ψηφιακών συστημάτων είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν και οι πολιτικές ομάδες λοιπόν έχουν καταλήξει σε μια συνένεση για να υπάρξει μια ερώτηση προς την Κομισιόν και ένα ψήφισμα για τα θέματα αυτά. Δίνω λοιπόν το λόγο στους εκπροσώπους. Ο κύριος Χιέλνερ είναι ο αρμόδιος για το ΕΛΚ, αλλά δεν είναι παρόν. Α, κύριε Βίνκλερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, ο Κρίστοφερ δεν είναι εδώ, είναι, δεν είναι προσωπική η ε, παρέμβαση, αλλά είναι το, η θέση του ΕΛΚ για το θέμα αυτό. Ε, θα σας παρουσιάσω λοιπόν τις, τα σημειώσεις του συναδέλφου Φιέλνερ. Νωρίτερα είδαμε την ολοκλήρωση όσον αφορά την, ανάθεση ε, εξουσιών μέσω του Omnibus. Πριν από αυτή την ολοκλήρωση το ε, σύστημα ήταν εξαιρετικά ξεπερασμένο και χρειάζονται ενημέρωση. Ένα από τα συμπεράσματα ήταν μια κοινή δήλωση και δύο δηλώσεις της Κομισιόν που ρητά ε, εξέφραζαν την ανησυχία της Κομισιόν όσον αφορά τα, ε, τις τεχνολογίες εποπτείας. Ε, σύγκληση των εξαγωγικών ελέγχων καθώς και η συμπερίληψη του μηχανισμού ε, ελέγχου. Εμεί τώρα αναμένουμε την Κομισιόν για να μας παρουσιάσει την πρότασή του στη πρότασή της για τον έλεγχο. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει αφού το εξετάσουμε. Δίνω το λόγο στον κύριο Λάιφρυντ, ο οποίο είναι διτή χρήση, λέει ο πρόεδρο. <laughs> Καλό είναι να έχω φίλου από την Επιτροπή, λέει ο κύριο Λάιφρυντ. Σα ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Δεν είναι δικό μου χόμπι το θέμα της διτής χρήσης, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και μόνη η δυνατότητα ορισμού του τι μπορεί να είναι διτής χρήσης και τι όχι είναι ένα δύσκολο πρόβλημα και το είδαμε αυτό στην τελευταία θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν είναι μονάχα τα υλικά αγαθά, ακόμα και το λογισμικό παρακολούθησης μπορεί να έχει διτό χαρακτήρα και όπως είπε και ο Πρόεδρός μας αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ε, Αραβικής Άνοιξης για να συλληφθούν αντιφρονούντες υπάρχουν ε, όμως διάφορα προϊόντα που έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά κάνουν πάρα πολύ δύσκολη την κατάσταση και είναι γνωστό ότι στο μέλλον θα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν στα κράτη-μέλη μας. Αυτό δεν είναι μονάχα δυσχερές, αλλά δημιουργεί και μια μεγάλη ανισότητα. Γι' αυτό εμεί θέλουμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν και πάλι να κάνει κάτι, γιατί εγώ προσωπικά είμαι απόλυτα δυσαρεστημένο για την καθυστέρηση τη πρόταση Κομισιόν, το γεγονό ότι γίνονται εξαγωγέ προϊόντων χωρί να υπάρχει πραγματικό έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε μονάχα κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχει καταχρηστική χρήση αυτών των προϊόντων και άμα η Κομισιόν δεν λέει απολύτω τίποτα για όλα αυτά, δεν είναι ικανοποιητικό αυτό. Περιμένω λοιπόν από την Κομισιόν να αντιμετωπίσει τα τρία ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει και θα ήθελα τώρα να ξέρω αν η Κομισιόν μπορεί να μας δώσει μια απάντηση και κυρίως πότε μπορούμε να περιμένουμε μια πρόταση από την Κομισιόν για να υπάρχει ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά γιατί νομίζω ότι είναι πια καιρό να γίνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Η Έμα. Το ECR ανησυχεί γιατί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα της διετής χρήσης και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι τεχνολογίες που έχουμε σήμερα μας προσφέρουν πολλά πλανεκτήματα και ευκαιρίες, αλλά υπάρχουν και τεράστιοι δυνητικοί κίνδυνοι σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν αυτές τις τεχνολογίες και γι' αυτό και η συμφωνία αυτή είναι μια ένα εξαιρετικό μέσο Και γι' αυτό και οι χώρες που παρέχουν ε, την έχουν υπογράψει. Και αυτό θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τους πιθανούς κινδύνους από την ακατάλληλη χρήση της τεχνολογίας, αλλά όμως θα πρέπει να παίζουμε σε ισότιμο πεδίο όσον αφορά τις ε, τεχνολογίες αυτές, γιατί περισσότερε ε, χρήσει είναι θεμητέ και πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ισότιμο πεδίο για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα εθνικά κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσουν την ασφάλειά τους. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι όλοι οι φορείς θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στη ε, διαδικασία αυτή, γιατί είναι πολύ τεχνικός, τεχνικό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται οι ε, έλεγχοι με τον κατάλληλο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το μέλη των υπόλοιπων ομάδων για τη συνεργασία τους. Αναφέρατε ότι εστιάζουμε στο θέμα και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε αυτό γιατί συνεχίζουν να αναπτύσσονται τεχνολογίες με πιθανό αντίκτυπο ανεπιθύμητο. Αυτό όλα έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων στις τρίτες χώρες και θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως boomerang και να χρησιμοποιηθούν εναντίον της δικής μας σημαντικής υποδομής και στρατηγικών συμφερόντων. Ε, πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν με δυνατότητες αναχέτησης αλλά και μέσω των ε, δυνάμων ε, των αστυνομικών εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς σε χώρες όπου δεν επικρατεί κράτος δικαίου. Αυτό είναι σημαντικό που τα κρατημέλη αναγνώρισαν ότι ο στρατηγικός αντίκτυπος είναι μεγάλος, που ενημέρωσαν τις ρυθμίσεις ε, ωστόσο δεν καλύπτονται όλες οι ανησυχίες που έχουμε από την ε, ρύθμιση Γι' αυτό και είναι κομμάτι της προφορικής μας ερώτησης. Θα θέλαμε η Κομισιόν να είναι πιο αποτελεσματική και να προβεί σε ενημερώσεις ε, που θα αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα θέματα και όπως είπε η συνάδελφος Κλάρκ είναι σωστό να υπάρχει ισότιμο πεδίο σε ολόκληρη την Ευρώπη γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξει αγώνας προς τα κάτω προς την μείωση των προδιαγραφών. Γιατί θα πρέπει οι κανόνες να είναι σαφείς και αυτό το ακούμε και από τις επιχειρήσεις και χρειάζεται η τεχνική πυρογνώμονε να μας ενημερώνουν διαρκώς για τον πιθανό αντίκτυπο όλων αυτών των ε, ε, τεχνολογιών. Πολύ σημαντική διαδικασία γιατί μπορεί να είμαστε μπροστά στην εκτίμηση του τι αντίκτυπο μπορούν να έχουν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι τεχνολογίες ε, ε, μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα στατικικά μας συμφέροντα, ενώ δεν υπάρχει προστασία, υπάρχει ένα κενό ε, ρύθμισης και εγώ ποτέ δεν είμαι υπέρ της υπερβολικής νομοθεσίας, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ ενημέροι όσον αφορά τους ελέγχους των εξαγωγών. Αυτή είναι η ουσία αυτή τη προφορική ερώτηση και νομίζω θα πρέπει να θεωρηθεί και ω ενθάρρυνση, ω παρότρινση παρότριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Μάλιστα, όντως. Ο Χέλμουντ Scholz. Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα θέματα αυτά ήταν αντικείμενο συζήτηση με πολλές ε, πολιτικές ομάδες και θέλω να τις ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ο εκ των προτέρων έλεγχος για τα προϊόντα διτή χρήση. Γιατί τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα, να είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν καταλήξουν σε λάθο χώρε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν, να μπορούμε να ξέρουμε τι δίνουμε σε τέτοιε χώρε. Αυτό δεν αφορά μόνο την αγορά αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικού στόχου, αλλά και για τεχνολογίε. Επίση, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτών των προϊόντων πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάζονται από ουδέτερους ερευνητές και ΜΚΟ με την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εμπορικά συμφέροντα είναι προφανώς μεροληπτικές και δεν πρέπει να έχουν αυτές τον αποφασιστικό ρόλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Φρανσίσκα Κέλλερ για τους πράσινους αλλά δεν τη βλέπω. Ε, κύριε Μπόμαν, όχι και για την ομάδα της ε, EFTD δεν έχω κανένα εισηγητή, σκιώδη. Δεν βλέπω κανέναν να θέλει να λάβει το λόγο, οπότε μπορώ να δώσω και πάλι στην Κομισιόν τον λόγο. Και στον κύριο Ασκουνίζε. Χαίρομαι που βλέπω ότι οι περισσότεροι δέχεστε τα στοιχεία της ανακοίνωσής μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τα σχόλιά σας και σημειώνουμε και τις ανησυχίες σας. Βέβαια πρόκειται για μια μακρά και δύσκολη διαδικασία. Ακόμη την εξετάζουμε και βουλευόμαστε τους ενδιαφερόμενους. Θα σας στηρίσουμε ενήμερους και για την περάτωση της διαδικασίας αυτής. Ευχαριστώ. Δεν σας κατάλαβα πολύ καλά για να με Εγώ νόμιζα ότι θα μου πείτε σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι προετοιμασίες της Κομισιόν για τη νέα νομοθετική ρύθμιση και πώς θα απαντούσατε στα τρία ερωτήματα που έθεσαν οι βουλευτές της Επιτροπής μας. Yeah, uh, can... Α, ναι. Μπορώ να σας πω ποια είναι τα τελευταία βήματα που έγιναν. Ένα βήμα βιομηχάνων στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες οργανώθηκε με εκπροσώπους της βιομηχανίας και εθνικούς εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Και εκεί διαβάσαμε μαζί την ανακοίνωση, συζητήσαμε τις τέσσερις προτεραιότητες που θέτει και πήραμε μερικές πληροφορίες από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Και βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό, είναι και πολιτικό και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβουν όλοι και να συμφωνήσουν επί των προτεραιοτήτων. Αλλά θα επανέλθουμε και θα σας πληροφορήσουμε στην επόμενη ευκαιρία με πιο ακριβή χρονοδιαγράμματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος η κυρία Σά και η κυρία Μακλάρεν σας έχουν ζητήσει να πείτε ποιο είναι το συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο θα έχει η πρόταση της Κομισιόν. Τι θα πει σε λίγου μήνε. αυτό δεν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο όταν λέτε. Εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτά που ακούσαν. Ο κύριο ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν. Μίλησε για δύο λεπτά και δεν είπε Νίξ δεν είπε τίποτα. Δεν θέλω να έχω εκπροσώπους της Κομισιόν οι οποίοι δεν απαντούν στα ερωτήματά μας. Αν είναι κάποιος που εκπροσωπεί την Κομισιόν θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Αυτή η κατάσταση είναι παράλογη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία αυτή να σας δώσω περαιτέρω λεπτομέρειες. Ούτως ή άλλως θέλω να σας καθησυχάσω η απάντηση στο ερώτημα στα ερωτήματά σας θα δοθεί στην Ολομέλεια. Έτσι δεν γίνεται πάντοτε. Αυτό δεν προδικάζει καθόλου τη δυνατότητα του Επιτρόπου να δώσει την απάντηση που αναμένεται. Καθόλου, στην Ολομέλεια. Ούτως ή άλλως όμως έτσι για να σας καθησυχάσω προετοιμάζουμε πολύ εντατικά την εξέταση της πρότασης και πολλοί συνάδελφοί σας είπαν ότι τα θέματα, οι μερικά θέματα είναι λεπτά και χρειάζονται αξιολόγηση και τεχνική ανάλυση. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα σας χορηγηθούν από την Επίτροπο Μάλστρομ όταν θα απαντήσετε... το προφορικό σας ερώτημα στην Αλαμέλεια. Μα θα έπρεπε να είσαστε στη διπλωματική υπηρεσία έτσι ωραία που τα λέτε, τόσο ευγενικά που τα λέτε. Αλλά δεν έχουν καμία ουσία όλα αυτά που λέτε, την οποία εμείς απαιτούμε από σας. Η δική μου πρόταση προς εσάς είναι στην επόμενη συζήτηση να έρθετε καλύτερα προετοιμασμένοι σε επίπεδο ουσίας και να είστε σε θέση να απαντήσετε. Ακόμα και στην Ολομέλεια είναι εκεί που θα πρέπει να υπάρξει η επίσημη απάντηση από την πλευρά της Κομισιόν, αλλά το νόημα της συζήτησης μαζί σας θα πρέπει να είναι να παίρνουμε πληροφορίες ουσίας και όχι απλώς να περιορίσετε σε διπλωματικές υπεκφυγές αλλά να συζητάμε σε επίπεδο ουσίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης, το σημείο υπαριθμών 9. Λοιπόν, σημείο 9. Πρόκειται για την κατάσταση που αφορά τους δασμούς για τα προϊόντα που προέρχονται από το Εκουαδόρ. Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι το Εκουαδόρ θέλει να συμμετάσχει στην εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και το Περού και επομένως υπάρχει και η ανάγκη να σκεφτούμε για τον περιφερειακό χαρακτήρα αυτή της ε, συμφωνίας. Έκλεισαν οι διαπραγματεύσει 17 Ιουλίου με το Περού και την, Κολο... την Κολομβία. Ξέρετε όλοι ότι οι διαπραγματεύσει, η διαδικασία της προσχώρηση μια χώρας σε μια συμφωνία χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Ξέρετε πολύ καλά τι έγινε στην περίπτωση της συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού Καταλαβαίνετε ότι από τεχνική έποψη τα πράγματα αυτά είναι δύσκολα. Υπάρχουν πολλά εμπόδια στο δρόμο. Για το Εκουαδόρ πρόκειται από την 1η Ιανουαρίου 2015 να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν πια οι πρόνοιες των γενικευμένων προτιμήσεων συν και επομένως θα δημιουργηθεί ένα χάσμα σε σχέση με τις ρυθμίσεις αυτές. Η πρόταση είναι λοιπόν να παρατείνουμε ε, το τωρινό καθεστώς μέχρι ότου μπορέσει το Εκουαδόρ να προσχωρήσει τη συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την Κολομβία και το Περού. Ο Χέλμουντ Σόλτ είναι ο μόνιμο συγγητή μα για το θέμα αυτό και θα του δώσω το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή δεν είδα ακόμη τον αρμόδιο από την Κομισιόν, θα περιοριστώ μόνο λέγοντας ότι φυσικά αρχίσαμε την επεξεργασία του σημαντικότατου αυτού κανονισμού πριν καταλήξει η διαδικασία της έγκρισης και εφαρμοστεί ο κανονισμός. Αλλά όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αλλάξει τους κανόνες των γενικευμένων προτιμήσεων έτσι ώστε οι χώρες με χαμηλά και μέσα εισοδήματα να μην συμμετέχουν πλέον στο πρόγραμμα αυτό. Ανάλογα με την οικονομική της ανάπτυξη μια χώρα δηλαδή μπορεί να τιμωρηθεί και αυτό πρέπει, σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε πολλοί συνάδελφοι και από την προηγούμενη θητεία αλλά και από αυτήν έθελσαν να θέσουν το θέμα αυτό για τον Ισημερινό αλλά Ίσως μερικοί συνάδελφοι θεωρούσαν ότι θα πιεστεί η κυβέρνηση του Ισημερινού για να μπει στην νέα αυτή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών αλλά ότι αναγνωρίζω πλήρως και συμφωνώ με το ότι ο Ισημερινός πήρε την απόφαση αυτή. Βέβαια το θέμα αφορά την ίδια τη χώρα και τις πολιτικές συζητήσεις και αγώνες που γίνονται εκεί ή που θα γίνουν η Κομισιόν προτείνει τώρα ένα κανονισμό ώστε να παραταθεί το καθεστώς το προτιμησιακό του GSP συν για το Εκουαδόρ ως μια προσωρινή λύση για το χρονικό διάστημα μέχρι ότου φτάσουμε στη Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου όπως είπατε προηγουμένως. Για τους πολίτες του Εκουαδόρ εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση και ζητώ από όλες τις πολιτικές ομάδες να συμφωνήσουν το ταχύτερο δυνατό να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για αυτόν τον κανονισμό, ώστε να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα χρονικά διαστήματα στα οποία το, κατά διάρκεια των οποίων το Εκουαδόρ θα μείνει εκτός του νυμφώνα του GSPC. Και χωρίς αυτό τον κανονισμό το Εκουαδόρ θα χάσει από 120 με 160 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αν λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτή τη χρονική πίεση και επειδή πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική μας, το δημοκρατικό μας καθήκον να βοηθήσουμε τους πολίτες του Εκουαδόρ, εγώ θέλω να προσκαλέσω τους σχεδοσυσιητές την επόμενη εβδομάδα να αναζητήσουμε μια συμβαστική λύση για τα θέματα αυτά. Οι αλλαγές τις οποίες εγώ προτείνω στον κανονισμό είναι περιορισμένες. <clears throat> Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι έχουν μεγάλη σημασία από την οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ε, προτείνω να αναφέρετε το δικαίωμα του Εκουαδόρ να εφαρμόζει μέτρα διαφύλαξης επί τη βάση των συμφωνιών διαφύλαξης του ΠΟΕ σε περιπτώσεις λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα για τους πολίτες του Εκουαδόρ και επίσης θέλω η Κομισιόν να πληροφορήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνεχιζόμενη συμμόρφωση του Εκουαδόρ με τις ε, ε, πρόνοιες που ισχύουν για όλες τις χώρες που είναι στο καθεστώς GSP συν, γενικευμένες προτιμήσεις συν. Ελπίζω λοιπόν ότι το Κομισιόν δεν θα υποστεί μεγάλο άχθος για την παράδοση αναφορών και επομένως η τροπολογία μου λέει ότι μπορούμε να δεχτούμε ένα απλώς βαθμολόγιο από την πλευρά του Εκουαδόρ ως αναφορά. Και επίσης η Κομισιόν πιστεύω δεν θα πρέπει να αναφέρεται ε, εκπεφρασμένα στον κανονισμό αυτό ώστε να μην βρεθεί ενώπιον κινδύνων να υπάρξουν ε, διαμφισβητήσεις από τον ΠΟΕ για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η έγκριση του κανονισμού χωρίς διαφυσβήτηση. Ένα στοιχείο όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτό χωρίς να θίξει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμά μας να έχουμε αρνησή κυρία για οποιαδήποτε πρόταση της Κομισιόν να ανασταλεί το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων. Επομένως ζητώ να μην γίνει δεκτή η δυνατότητα της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει μια εφαρμοστική πράξη τον κανονισμό αυτό για τη γενικευμένη προσέγγιση και πρέπει η Κομισιόν να παραμείνει πιστή με το συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται αυτές οι ε, ρυθμίσεις. Και εμείς θα πρέπει στον ευρωπαϊκό δίκαιο να κρατήσουμε προβλέψιμη τη στάση μας. Δεν θέλουμε η, προϊόν, παραγωγή προϊόντος στο Εκουαδόρ να αντιμετωπίσουν από τη μια μέρα στην άλλη μια ριζική αλλαγή. Θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν και τις δημοκρατικές μας διαδικασίες και γι' αυτό θα ήθελα τέλος να σας αναφέρω και δύο περαιτέρω τροπολογίε που θέλω να καταθέσω αφορούν τα στοιχεία της αιτιολογικής σκέψης 6 που αναφέρεται στο άρθρο 3β. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για μέτρα από τον κατάλογο των στοιχείων που θα μείνουν εκεί. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει εκεί μια αλλαγή και στα αγγλικά θέλω να τροποποιήσω ορισμένες τη λέξη αυτή για τα μέτρα που δεν είναι πρέπουσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω αγαπητοί συνάδελφοι για τη συνεργασία σας σε σχέση με το θέμα αυτό και σας προσκαλώ να συνεχίσετε με το πνεύμα αυτό για να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία προς το συμφέρον των πολιτών του Εκουαδόλ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσβλέπω στις ε, παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος και ο Σχίζατς. Φύσας, ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, πρώτα απ' όλα Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτς για το έργο του και να σας πω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Έχουμε εξετάσει από κοινού όλα αυτά τα ζητήματα. Και επομένω, όπω ελέγχθη προηγουμένω, εμεί υποστηρίζουμε απόλυτα και χαιρετίζουμε την πρόταση κανονισμού η οποία θα επιτρέψει την παράταση των δασμολογικών προτιμήσεων για το Εκουαδόρ για το σύστημα μέχρι ότου τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, <clears throat> αλλά πιστεύω ότι είναι επαρκές ώστε ο κανονισμός αυτός να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί από την Κομισιόν και δεν θα εισαγάγουμε καμία τροπολογία σχετικά, όπως είπε ο κ. Σόλτς ως εισηγητής. Έχει ήδη ο ίδιος παρουσιάσει ορισμένε τροπολογίες, κάποιες από τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε, άλλες δεν Έχουμε, κάποιες, έχουμε αντίρρηση για αυτές, αλλά έχουμε κάποιες αμφιβολίες και πρέπει να τις αναλύσουμε περισσότερο. Η τροπολογία 5 <clears throat> που αφορούν το σημείο 6 του άρθρου 3β σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του Εκουαδόρ να εφαρμόσει μέτρα διαφύλαξης. Φυσικά έχει το δικαίωμα αυτό το Εκουαδόρ. Ίσως όμως να είναι υπερβολικό να υπογραμμίζεται αυτό το σημείο. Εγώ δεν βλέπω πρόβλημα για αυτές τις τροπολογίες από την ομάδα μας. Για τις τροπολογίες τώρα 2, 4 και 6. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση των αιτιολογικών σκέψεων 7, 10 και του άρθρου 3 και βάζουμε μια σύνδεση με τον κανονισμό GSP. Εγώ συμφωνώ επί της σε ενοιολογικό επίπεδο, αλλά έχω κάποιε ε, αμφιβολίες, γιατί ενδεχομένως αυτή η σύνδεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικά προβλήματα. Πριν λοιπόν υποστηρίξω αυτές τις τροπολογίες, θα ήθελα να έχω την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει κάποια ε, προσφυγή στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σε σχέση με την νομιμότητα αυτής της ρύθμισης. Υπάρχει τώρα η τροπολογία 3 για ένα νέο μια νέα αιτιολογική σκέψη 9α ώστε η Κομισιόν να πληροφορήσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το νέο κανονισμό και συμφωνούμε απόλυτα για τι τροπολογίε 4, 7, 8, 9 και 10 θα έχουν σαν αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η αιτιολογική σκέψη 10 και το σημείο 4 και λένε ότι θα πρέπει να γίνει με κατεξουσιοδότηση πράξη η άρση του συστήματος γενικευμένων ε, προτιμήσεων και όχι με μια εκτελεστική πράξη όπως ζητάει η Κομισιόν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύπλοκο λόγω του περιορισμένου στο χρόνο χαρακτήρα αυτού του κανονισμού ίσως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όπως ζητάει ο εισηγητής. Από τη στιγμή που ξεκινάει η Κομισιόν τη διαδικασία της προσωρινής άρσης του συστήματος γενικευμένων προς ε, προτιμήσεων μέχρι να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο μπορεί να περάσει 1,5 έτος και στην περίπτωση του κανονισμού που μας ενδιαφέρουν αυτό ουσιαστικά δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια χρονική άρση των προτιμήσεων του προμηθυσιακού συστήματος. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που είναι πιο ευέλικτο και πιο γρήγορο από αυτό το οποίο προβλέπει ο κανονισμός. Και από την άποψη αυτή ξέρω ότι ζητήθηκε από τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφράσουν γνώμη για το αν πρέπει να είναι κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξει αυτέ οι οποίε θα εφαρμοστούν. Γι' αυτό πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να περιμένουμε τη γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία. Και φυσικά παραμένω στη διάθεση του εισηγητή και όλων των σκηριωδών εισηγητών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και να καταλήξουμε στη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Και ούτω ή άλλω ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αίσιο πέρα σε σχέση με την διαπραγμάτευση αυτή για να μην υπάρξουν προβλήματα τα οποία μπορούν να γίνουν για τους εξαγωγείς του Εκουαδόρ ή τους εισαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η... Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Φίσας εγώ ως εισηγητής για τους σοσιαλιστές θα πω ότι έχουμε τρεις προκλήσεις ενώπιόν μας με το προτινόμενο νομοθέτημα. Πρώτα απ' όλα, πρώτα θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι από τη στιγμή που θα εκπνεύσει ο κανονισμός και από, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία η εμπορική δεν πρέπει να υπάρχει ένα κενό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στον 1,5 χρόνο, γιατί μπορεί η διαδικασία κύρωσης να καθυστερήσει περισσότερο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε την απαραίτητη ευκαμψία στα θέματα αυτά. Σε 1,5 χρόνο θα έχουμε ήδη το ίδιο πρόβλημα, εάν δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης. Δεύτερον, η δεύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι επί τη βάση αυτών των προτιμήσεων οι υποχρεώσεις που συνάπτονται με το καθεστώς των γενικευμένων προτιμήσεων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Δηλαδή να υπάρξει η νομική αυτή δέσμευση. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτό. Από τη μία πλευρά μπορούμε να πούμε ότι παραμένουν αυτές οι υποχρεώσεις και η εποπτεία τους. Ο άλλος τρόπος θα ήταν να ζητήσουμε και στο μεταβατικό διάστημα να εφαρμοστούν οι πρόνοιες της συμφωνίας που εμπλέκει την Κολομβία, το Περού και στο μέλλον και το Εκουαδόρ ή τουλάχιστον να εισαχθούν σταδιακά. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι για τα θέματα της αηφορίας θα πρέπει να εφαρμοστεί, να εφαρμόσει το Εκουαδόρ στην ε, περίπτωση στο διάστημα αυτό της ε, ε, μεταβατικής περίοδου μέχρι την ανάληψη της συμφωνίας. Το στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε βέβαια την διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι τα δικαιώματά μας με την μεταφορά από πράξεις κατά σε εκτελεστικές πράξεις δεν διατηρούνται. Γι' αυτό από λόγους ε, ουσίας και λόγους αρχής πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις αλλά έχετε δίκιο, είναι καλό να έχουμε από τη νομική υπηρεσία μια γραμμοδότηση την οποία θα συζητήσουμε μεταξύ των συντονιστών. Αλλά και αυτό θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο που θα λάβουμε υπόψη εγκαίρως. Αυτά λοιπόν ως σκιώδης εισηγητής από τους σοσιαλιστές. Τώρα ξαναβάζω το κασκέτο του Προέδρου και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο σκιώδη εισηγητή από τους συντηρητικούς. Δεν βλέπω να είναι παρόν όμως. Η Μαρίκε από τους φιλελεύθερους έχει το λόγο. Η Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εξ ονόματος Ρεμόν Τρεμός που είναι ο σκιώδης μας. Η ομάδα μας είναι υπέρ που συνόλου τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Κολομβία. Η συμφωνία του Ιουλίου μεταξύ Ένωσης και Ισημερινού είναι ένα βήμα περαιτέρω για περισσότερη πρόσβαση στις αγορές μας και αυτό είναι θετικό. Βέβαια είναι μικρή αγορά ο Ισημερινός αλλά υπάρχουν ορισμένοι συγκεκριμένοι τομείς που έχουν αναπτυξιακό δυναμικό προτείνει η Κομισιόν να παραταθούν, να επεκταθούν οι προτιμήσεις και πέρα από το Δεκέμβριο 14 μέχρι να αρχίσει να ισχύει, να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία αυτή, όπως λέει και ο εισηγητής, δεν θα καθυστερήσει χωρίς λόγο και με αυτόν τον, τον στόχο θα, με αυτόν τον στόχο εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα αξιολογήσουμε και την άποψη της νομικής υπηρεσίας ως προς την συνέπειά του κειμένου αυτού με άλλες συμφωνίες. Ελπίζουμε ο Ισημερινός να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να μπορέσει να στηρίξει τη δημιουργία ενός θετικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Ο κύριος Μποβέ δεν είναι παρόν. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν. Ποιος θα ήθελε, κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να παραστούμε και εμείς σήμερα σε αυτή τη συνάντηση. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το Κοινοβούλιο διεκπεραιώνει γρήγορα αυτό το θέμα και περιμένουμε να δούμε τι προτάσεις θα κάνετε για τροπολογίες και μετά μπορώ να σας πω ότι θα συμμετάσχουμε επικοδομητικά στη διαδικασία γενικότερης διεκπαιρέωσης μέσα στην νομοθετική διαδικασία δηλαδή από τους δύο συνομοθέτες ελπίζουμε χωρίς καθυστερήσεις και αν χρειαστεί θα διευκολύνουμε την εργασία τους αν χρειαστούν τίποτε προσαρμογές, τίποτε άλλες αλλαγές που θα ζητήσουν οι συνομοθέτε. Παρ' όλα αυτά, η πρότασή μας και για το θέμα των εφαρμοστικών πράξεων και των τι αυτών ή ούτων. ε, στηρίζεται στα επιχειρήματα που αναφέραμε γραπτός. Αλλά προς το παρόν επαναλαμβάνω περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις και τροπολογίες. Σας ευχαριστώ το θέμα του χρονικού περιεχομένου, του χρονικού ορίου. Είσαστε σίγουρος ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι επαρκής για να καλύψει τα θέματα της κύρωσης. Ναι, πράγματι πιστεύουμε ότι αν προχωρήσουμε με τον σωστό τρόπο και υπάρχει η φυσιολογική χρονική αλληλουχία και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα σε δύο χρόνια θα μπορούμε να έχουμε περατώσει αυτή τη διαδικασία. Για το Πέρου και την Κολομβία χρειάστηκε λίγο παραπάνω από δύο χρόνια από το τέλος των διαπραγματεύσεων για να τεθούν σε εφαρμογή, αλλά ήταν και πιο πολύπλοκη νομική κατάσταση. Και υπήρχαν και κάποια ουσιοδέστερα πολιτικά προβλήματα που έπρεπε να επιληθούν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπήρχαν και θέματα εφαρμογής που είχαν να κάνουν με τη γεωγραφική ένδειξη προέλευσης. Όλα αυτά χρειάστηκαν πιο πολύ χρόνο στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξαν κάποια πολιτικά θέματα. Η ελπίδα μας είναι ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα θέματα αυτά στην περίπτωση του Εκουαδόρ. Αλλά ας το δούμε στο δρόμο. Εμείς πιστεύουμε ότι φτάνει ο χρόνος. Εντάξει, ο κύριος Σάιβα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια σε ό,τι αφορά την εργασία μας και την επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Περού και την Κολομβία και μετά θέλω να επανέλθω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος μου ο και οι άλλοι συνάδελφοι για τη συμφωνία του να έχουμε την ε, ε, ρύθμιση αυτή ώστε οι εξαγωγές του Εκουαδόρ να μην βρεθούν εκτός του καθεστώτος αυτού γενικευμένων προστιμήσεων. Και επίσης να μην υπάρξει και Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Επιμένουμε λοιπόν και πάλι ότι φυσικά θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά το νομικό επίπεδο, ώστε να μην διαμφισβητηθεί αυτή η συμφωνία ω αντιτιθέμενη στου κανόνε του ΠΟΕ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι εισηγητέ και οι ισχυρότερε εισηγητέ θα κάνουν όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορέσουν να διασκεδαστούν όλε αυτέ τι νομικέ ανησυχίες. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κάποιο άλλο θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Επανέρχομαι και πάλι στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο για τα σχόλιά τους. Έχω μιλήσει και με πολλούς από αυτούς ήδη. Έχω λάβει και, όπως είπα και προηγουμένως, και με μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Θέλω να σας παραπέμψω τώρα σε τέσσερα βασικά σημεία ε, θέματα. Υπάρχουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον κανονισμό για τις γενικευμένες προτιμήσεις. Χρειάστηκε λοιπόν να καταδαπανίσουμε πολύ χρόνο για να καταλάβουμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βρίσκονται τα δικαιώματα εποπτείας του νομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πότε λοιπόν μπορούν να αρθούν οι προτιμήσεις ή καλύτερα πότε μπορούν να αρθούν συγκεκριμένες ρήτρε που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία για τις γενικευμένες προτιμήσεις. Και αυτό το λέω στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν αμφιβολία γιατί, για το αν εμείς πρέπει να διατηρήσουμε τα δικαιώματά μας σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για χρονικό ορίζοντα σε ό,τι αφορά αυτή την νομοθεσία. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω, το ζήτημα της εποπτείας. Είχαμε μια συνάντηση και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία και τη θέληση να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα έχουν γνώση των λόγων για τους οποίους εμείς έχουμε κάνει αυτή την πρόταση. Είχα επίσης την ευκαιρία να μιλήσω με τον Υπουργό Εμπορίου της Δημοκρατίας του Ισημερινού την προηγούμενη εβδομάδα, του Εκουαδόρ, και ο οποίος και πάλι μου επέσε την προσοχή ότι όλα αυτά κυρίως είναι απαραίτητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Εκουαδόρ, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με την θέση σε εφαρμογή της Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περού καθώς και της Κολομβίας και οι οποίοι τίθενται ενώπιον ενός δύσκολου πλαισίου. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο. Καλά είναι να μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά όλα αυτά τα οποία λέμε έχουν και πραγματικές συνέπειες για τις συνθήκες εργασίας πάρα πολλών ανθρώπων στο Εκουαδόρ. και η σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ του Περού και της ε, Κολομβίας έχει οδηγήσει σε μείωση σημαντική των εσόδων αυτών των ε, επιχειρήσεων και των εργαζομένων στο Εκουαδόρ. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους ε, εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σε σχέση με τη συμβατότητα όλων αυτών με τους κανόνες του ΠΟΕ. Και γι' αυτό τονίζω ότι θα πρέπει εκ των προτέρων να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ελέγξουμε κατά πόσο συνάδουν όλες αυτές οι ρυθμίσεις με το δίκαιο του ΠΟΕ. Χαίρομαι λοιπόν για τη δυνατότητα να έχουμε μια καλή συνεργασία Προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητές και ελπίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο το οποίο μπορεί να ε, συμπεριλάβει τις τροπολογίες των ώστε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο σφιχτό χρονοδιάγραμμα που έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας να μπορέσουμε να φέρουμε σε τέλος, σε αίσιο Να μπορέσουμε λοιπόν να συμπληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ για την πλήρη αυτή παρουσίασή σας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την εξέταση αυτού του θέματος. Κλείνει λοιπόν και αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και το πρώτο τμήμα της ημερησίας διάταξής μας ε, και στις 11 η ώρα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ε, 11 o'clock λέω Σας ευχαριστώ.